Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να προσπαθήσετε να καθίσετε. Γιατί θα αρχίσουμε την ιδρυτική μας συνεδρίαση. Καθίστε παρακαλώ. αρχίσω. Γι' αυτό παρακαλώ καθίστε και η πίσω και η πίσω έχει θέσεις πίσω. Okay. So... Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλωσορίζω, σας καλωσορίζω εδώ ιδιαίτερα τα νέα μέλη της Επιτροπής μας θα προεδρεύσω μέχρι να εκλεγεί ο πρόεδρός μας. Άρχεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ όμως καθίστε. Σας υπενθυμίζω ποιος είναι ο στόχος της σημερινής μας συνάντησης να εκλέξουμε το Προεδρείο, δηλαδή τον Πρόεδρο και μέχρι τέσσερις αντιπροέδρους, σύμφωνα με τον κανονισμό το άρθρο 234. Πρώτα, 204. Πρώτα θα εκλεγεί ο Πρόεδρος. Παρακαλώ συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε γρήγορα γιατί σε λίγη ώρα θα έρθει και άλλη επιτροπή εδώ να εκλέξει. Λοιπόν, Παρακαλώ καθίστε. Λοιπόν, θα εκλέξουμε πρώτα τον Πρόεδρο και μετά τους Αντιπροέδρους. Σύμφωνα με το άρθρο 200 του κανονισμού, πρέπει να σας ανακοινώσω ότι οι ακόλουθοι αναπληρωματικοί συμμετέχουν αντί αναπληρώνοντας τα πλήρη μέλη για το ΕΛΚ Κοέλιο αντί του κυρίου Μπέκερ Τσάκη αντί για Χολμάγερ Μένες Μπέσερ Μπαριοτερέζα αντί για Ορτεφε κυρία Μωράνο αντί για την κυρία Μακοβέη κυρία Τούν αντί για την κυρία Ματέρα Βότσενμπεργκ αντί για Ματσόλα και Και Μουσολίνη αντί για Χολμάγερ, λάθος έκανα πριν. Ε, και ο κύριος Κύρκος αντί για την κυρία Φαγιόν, η κυρία Πύλη για την κυρία Φρασίκο Βαμπένοβα, κυρία Σλέιν για τον κύριο Λόπες Αγκυλάρ και για τους συντηρητικούς κύριος Τόμσιτς αντί του κύριου Κίρκοπ, Γιούρεκ αντί για Τόμασεύσκι, για τους ηλελεύθερους Ροσφόρ αντί για Φρίσμπακ, Παγκαζολτούντου αντί για Λουί Μισελ και μετά ξανά ψηφιδικούς Κάρσον αντί για Βιασδόνσκι. Spinelli Σπινέλη αντί για Άντερσον. Άλλη αλλαγή. Ο κύριος Λέναρτ αντί για τον κύριο Σόγκολ. Αυτά χρειάστηκε να σας τα ανακοινώσω. Αυτοί οι ανεπληρωματικοί μπορούν να ψηφίσουν στη θέση των πλήρων μελών που αντικαθιστούν. Τώρα, ως προς την απαρτία, χρειάζονται πάνω από 50 μέλη, νομίζω είναι παρόντα υπάρχει απαρτία. Χρειαζόμαστε 15 μέλη τουλάχιστον εδώ, ένα τέταρτο δηλαδή των 60 μελών. Άλλη αλλαγή, η κυρία Κιέγκα θα ψηφίσει αντί της κυρίας Ρεβόνταλόν. Μάλιστα. Τώρα οι υποψηφιότητες. Ποιοι είναι οι υποψήφοι για την Προεδρία, για τον Πρόεδρο. Λοιπόν, η υποψηφιότητα θα κατετεθεί είτε από πολιτική ομάδα είτε από τουλάχιστον 5% των μελών. Στην περίπτωσή μας δηλαδή τρία μέλη. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής και να έχει συμπληρώσει τη δήλωση δημοσιονομικών συμφερόντων του. Ποιοι είναι λοιπόν, ποιοι ορίζονται υποψήφοι. Κυρία Ζήμπκα. Προτείνω εξ των σοσιαλιστών τον Κλοντ Μωράης. Μάλιστα. Κλοντ Μωράης. Άλλοι υποψήφοι. Όχι. Τότε ο υποψήφιος συμφωνεί. Συμφωνεί. Συμφωνώ. Συμφωνεί. Ευχαριστώ Κλόντα. Λοιπόν, ο υποψήφιος έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ανέφερα καθώς και τη συμπλήρωση των δημοσιονομικών συμφερόντων, είναι πλήρες μέλος και αφού είναι μόνο ένας ο υποψήφιος λέω να γίνει διαβοής. Φαντάζομαι συμφωνείτε διαβοής. Λοιπόν, βοόμεν. Συγχαρητήρια κύριε Μωράες. Έχει εκλεγεί διαβοής ο υποψήφιος και τον παρακαλώ να καταλάβει την θέση του Προέδρου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριοι συνάδελφοι. First of all, thank uh, Σε ευχαριστώ Κίνγκα, ευχαριστώ συνάδελφοι για την τεράστια τιμή που μου κάνατε να εκλεγώ πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Πριν συνεχίσουμε για την εκλογή των αντιπροέδρων, που δεν θέλω να την καθυστερήσω, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι συγκινημένος που έγινα πρόεδρος της Επιτροπής μας Μερικοί από εσά ε, ήταν και παλαιότερα μέλη της Επιτροπής αυτής και με ξέρετε, γνωρίζετε όλοι ότι η Επιτροπή είναι από τις σπουδαιότερες του Κοινοβουλίου γιατί ασχολείται με θέματα αξιών. Αυτά τα παλαιά μέλη λοιπόν έχουν ασχοληθεί με μερικά από τα σημαντικότερα νομοθετήματα και θα ασχοληθούν με τα σημαντικότερα νομοθετήματα που θα αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο. Όχι μόνο την οικονομία αλλά και τις αξίες που αντιπροσωπεύουμε στην Επιτροπή Ελευθεριών Δικαιοσύνης, θέματα δηλαδή όπως η συμμεταχείριση, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μετανάστευση, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι λοιπόν τεράστια η τιμή και σας κατευχαριστώ γι' αυτό. Συνεχίζουμε τώρα στην εκλογή των αντιπροέδρων. Πρώτον, σύμφωνα με το άρθρο 204 του κανονισμού, ε, να ανακοινώσω τους αναπληρωματικούς που θα ψηφίσουν. Ο ίδιος κατάλογος είναι όπως και πριν, ακριβώς ο ίδιος. Α, ακριβώς ο ίδιος. οι πολιτικές ομάδες είναι υποχρεωμένες να πληροφορούν τον Προεδρεύοντα για οποιαδήποτε αλλαγή των αναπληρωματικών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Λοιπόν, αρχίζει η εκλογή των Αντιπροέδρων. Ως προς την απαρτία υπάρχουν πάνω από 15 μέλη, υπάρχει απαρτία. γιατί το 1 τέταρτο των 60 μελών είναι 15. Λοιπόν, υποψηφιότητες. Πρώτα για τον πρώτο αντιπρόεδρο. Τον πρώτο αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ΕΛΚ προτείνει την κυρία Κίνγκα Γκάλ ως πρώτη αντιπρόεδρο της Επιτροπής Λίμπε. Πρώτη υποψηφιότητα για πρώτο αντιπρόεδρο λοιπόν η κυρία Κίνγκα Γκάλ. Για δεύτερο αντιπρόεδρο εξ ονόματος των σοσιαλιστών προτείνω την κυρία Γιώτοβα για δεύτερη αντιπρόεδρο. Η Λιάννα Γιώτοβα λοιπόν. Και τρίτο αντιπρόεδρο, τρίτο, Σαρτζεντίνη. Οι πράσινοι προτείνουν τον κύριο Όλμπρεχτ για τρίτο αντιπρόεδρο. Γιάνν Φίλιπ Όλμπρεχτ. Τέταρτος αντιπρόεδρος. Εξ ονόματος του ΕΛΚ προτείνουμε την κυρία Μπάρβαρα Κούντριτσκα. Πάει και ο τέταρτος υποψήφιος λοιπόν για τέταρτο αντιπρόεδρο οι υποψήφοι δέχονται την υποψηφιότητά τους. Όλοι, μάλιστα. Μάλιστα. Άλμπρεχτ, Ιώτοβα, Κιγκαγκάλ. Όλοι, όλοι συμφωνείτε, μάλιστα. Κοντέτκα. Έχετε όλοι συμπληρώσει ελπίζω τις δηλώσεις για τα δημοσιονομικά συμφέροντα μάλιστα. Ωραία, ελάτε να καθίσετε τότε. Ή μάλλον όχι πρέπει να τα κάνουμε δημοκρατικά. Πριν έρθατε να καθίσετε, πριν έρθετε να καθίσετε, μην νομίζετε ότι παρέλειψα τους δημοκρατικούς κανόνες, πρέπει ή να ψηφίσουμε ή να το κάνουμε διαβοής. Λοιπόν, διαβοής. Ψηφίζουμε διαβοής. Τώρα οι αντιπρόεδροι παρακαλώ να έρθουν να καθίσουν. Okay, colleagues, um... Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς θερμά μας. Έχω ακόμα δύο διαδικαστικά. Την επικύρωση του προγράμματος εργασιών για το υπόλοιπο του χρόνου. Έχετε λάβει το σχέδιο και δεν θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν αντιρρήσεις όχι από ό,τι βλέπω. Α, η πρώτη αντίρρηση επί προεδρίας μου λοιπόν, κυρία Σαρσεντίνη. Ναι, ναι, είμαι υπερήφανη γι' αυτά. Δεν θα πω ότι είναι και αντίρρηση προεδρέα, αλλά θέλω να επισημάνω πως προβλέπονται δύο συνεδριάσεις που αρχίζουν πέμπτη απόγευμα 3 και τελειώνουν 6.30. 14 Σεπτεμβρίου η πρώτη και 6 Νοεμβρίου η δεύτερη. Ξέρετε πολύ καλά όπως και εγώ ότι οι συνεδριάσεις που πάνε μέχρι αργά το απόγευμα της Πέμπτης δεν στέφονται με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω εάν πράγματι πιστεύετε ότι θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις αυτές. Yeah. thank you for, um, helping. Ευχαριστώ πολύ που με βοηθάς αυτή την πρώτη συνεδρίαση στην οποία προεδρεύω. Αυτά οι συνημερομηνίε που μα έδωσε η διάσκεψη των Προέδρων. Και η διάσκεψη των Προέδρων έδωσε, η διάσκεψη των Προέδρων θα πάρει. Έτσι λοιπόν, προς το παρόν μένει αυτό. Θα το δούμε και με τους συντονιστέ. Ε, υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις για το πρόγραμμα. Μια και είσαστε όλοι καινούργοι στην συνεδρίαση θα εγείρω το θέμα και με τους συντονιστές και θα επανέλθουμε να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Δεύτερο θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν μου φύγετε. που έχει επίσης αποφασίσει τη σκέψη των Προέδρων, η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών θα δεχθεί σε ακρόαση τους, τον υποψήφιο στην υποψήφιο για θέματα δικαιοσύνης στις 14 Ιουλίου μαζί με την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων και των Δικαιωμάτων των Γυναικών, την κυρία Ρέντινγκ. Και η ψηφοφορία θα γίνει 5η 10 Ιουλίου. Ξέρετε ότι η κυρία Ρέντινγκ αντικαθίσταται και ως εκ τούτου πρέπει να ε, δούμε τον αντικαταστάτη τη. Γι' αυτό γίνεται αυτή η ακρόαση. Για να δούμε τον αντικαταστάτη τη, κυρία Γκρέτελ. Αντιρρήσει. Ωραία. Η προσεχής μας συνεδρίαση προβλέπεται για τι 14 Ιουλίου. Τίποτε άλλο στο διάφορο. Όχι. Ήμουν κάπως ε, συγκινημένος με την ευκαιρία αυτής τη εκλογής μου. Ζητώ συγγνώμη. Θέλω να πω πάντως για τους παλαιότερους συνάδελφους που με γνωρίζουν ήδη ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν και προς τους νέους συναδέλφους ότι θα είμαι πάντα δι... ακριβοδίκαιος απέναντι σε όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτω ομάδος. Έχουμε σημαντικά θέματα να συζητήσουμε στην Επιτροπή μας, δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα χρειαστεί να τα δούμε με μεγάλη υπομονή, με πολύ σκληρή δουλειά και βέβαια με πολύ καλή διάθεση. Λάθη θα κάνουμε, λάθη θα κάνω. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι όσο το δυνατόν πιο ακριβοδίκαιο στην Επιτροπή μου και στα καθήκοντά μου και ότι θα εργαστώ το δυνατόν πιο σκληρά αυτά τα δυόμιση χρόνια ή και πέντε αν με επανεκλέξετε στα μισά της θητείας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την εμπιστοσύνη σας και περιμένω να δουλέψουμε όλοι μαζί πολύ καλά.